με τη σειρά. Πρέπει να σας κάνω μια ανακοίνωση. Ο κύριος Βλάντιμιρ Ρέμεκ με ενημέρωσε ότι παρετείται από μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις 16 Δεκεμβρίου 2013 και με ενημέρωσε σχετικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού, διαπιστώνει τη χειρία της έδρας από τις 16 12 του 2013 και ενημερώνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές σχετικώς. Κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε λοιπόν στις ψηφοφορίες. Ο κύριος Μπρόκ ζητεί το λόγο για διαδικαστικό, για τον κανονισμό. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ενημερώσω το σώμα επειδή θα ψηφίσουμε για την Ουκρανία σε λίγο, ότι εδώ και τρεις ώρες η κόρη και ο συνήγορος της κυρίας Γιούλια Τιμοσέγκο δεν έχουν το δικαίωμα να την επισκεφθούν στη φυλακή. Τους έχει απαγορευτεί η είσοδος, είναι μπροστά στη φυλακή και παραβιάζοντας την νομοθεσία της χώρας δεν τους επιτρέπουν να επισκεφθούν την κυρία Τιμοσέγκο, η κόρη της και ο δικηγόρος. Ευχαριστώ ε, για την ανακοίνωση αυτή που είναι πολύ λυπηρή και δείχνει πόσο έχει κλιμακωθεί η κατάσταση στην Ουκρανία και πόσο σημαντική θα είναι η επόμενη διαδικασία και από